και στα πρακτικά της συνεδριάσεως αυτής. Θα ήθελα να σας πω ότι την Πέμπτη ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου θα ψηφίσει βάσει του άρθρου 74 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα υπογράψει, λέω, 12 πράξεις υπό την συνήθη νομοθετική διαδικασία. Κείμενα ε, και οι τίτλοι των πράξεων μάλλον θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα. Κύριε Μποργέτσιο, έχετε ζητήσει το λόγο επί του κανονισμού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, ναι. Σήμερα το πρωί στην Ελλάδα, στο Βένετο, 30 ε, άνθρωποι, 30 άτομα έχουν ε, ε, χωρίς κανένα πρόβλημα στο ποινικό τους μητρό έχουν συλληφθεί από την αστυνομία μόνο και μόνο γιατί διαδήλωναν <clears throat> υπέρ της ανεκδησίας του Βένετο. Πρόκειται για έγκλημα κατά της ελευθεροτυπίας και της ελευθερίας έκφρασης των ιδεών σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κύριε Μποργέτζιο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το θέμα είναι εντελώς άσχετο με την ημερήσια διάταξη. όλα αυτά καταγράφει η Προεδρία της δηλώσης σας. Κυρία Γκρέσλερ, παρακαλώ. Eine Kritik anzubringen an dem Herrn Parlamentspräsidenten, der im Bericht über die Parlamentsentlastung einen Paragraphen des Haushaltskontrollausschusses für unzulässig erklärt hat, und zwar den Paragraphen 47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 Λειτουργεί τώρα η διερμηνία πολύ ωραία. Οι παρατηρήσεις σας, κυρία Γκρέσλερ, οι οποίες σχετίζονται με την απαλλαγή, θα πρέπει να γίνουν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 η νομική βάση από ό,τι μου λένε οι αρμόδιοι είναι το άρθρο 20. Εν πάση περιπτώσει όμως ε, οι παρατηρήσεις σας αυτές θα πρέπει να γίνουν όταν θα ξεκινήσει η συζήτηση για το ε, ζήτημα της ημερησίας διάκτησης που θα ασχοληθεί με την απαλλαγή. Τώρα θα σας δώσω κάποιες πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση της ημερησίας διατάξεως. Όταν λοιπόν θα φτάσει η συζήτηση στο σημείο το οποίο ασχολείται με την απαλλαγή θα σας καλέσω να κάνετε τις σχετικές σας παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Περνούμε λοιπόν στην ημερήσια διάταξη όπως, ε, όπως ορίστηκε από, την, ε, από τους Προέδρους των ομάδων. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις τροποποίησης της ημερησίας διατάξεως. Τετάρτη 2 Απριλίου. Η κοινή συζήτηση για την